Αγαπητοί φίλοι, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους σας, τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και όλους τους υπόλοιπους από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, από το Πολωνικό Κοινοβούλιο, όλους ε, εκτός Ευρώπης, όλους όσους ήρθατε σήμερα εδώ. συνεδριάζουμε για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους 96 ανθρώπους που έχασαν τραγικά τη ζωή τους το Σάββατο στο Σμόλενξ. Μεταξύ αυτών, ένας πρόεδρος ενός ευρωπαϊκού κράτους και 18 βουλευτές. Οι συνάδελφοι από το Εθνικό Κοινοβούλιο, δημοκρατικά εκλεγμένοι από τον πολωνικό λαό. Οι σκέψεις μας, Χριστός, βρίσκονται κοντά στις οικογένειες και στους αγαπημένους ανθρώπους των θυμάτων. Τα μηνύματα στήριξης που έλαβα από τόσο πολύ κόσμο, τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, τους πρεσβευτές, τις διοικήσεις των ευρωπαϊκών οργανισμών, το προσωπικό, τους δημοσιογράφους, αλλά και ανθρώπους εκτός Ευρώπης, έδωσαν σε μένα και στη χώρα μου κάποια δύναμη και ανακούφιση. Το εκτιμώ πάρα πολύ αυτό. Και είμαι περήφανος. Μπορούμε όλοι να είμαστε περήφανοι για το πώς αντέδρασε το έθνος μας. Πρόκειται για μία άνευ προηγουμένου καταστροφή. Χάθηκαν υπηρετώντας τη χώρα τους στο δρόμο για την τελετή για εκείνους που έχασαν τη ζωή τους στο Κατίν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο η ιστορία με δραματικό τρόπο έκλεισε έναν πλήρη κύκλο. Μα συγκίνησε και η αντίδραση της Ρωσίας, που ήταν γεμάτη αξιοπρέπεια και κατανόηση. Ευχαριστώ τους Ρώσους φίλους μας. πιστεύω πως θα μας βοηθήσει ώστε να συμφιλιώσουμε την ήπειρό μας μέσα στο πλαίσιο της ιστορικής αλήθειας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού. Ξέρω πως η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της χώρας μου, της Πολωνίας. Σε αυτή τη τόσο δύσκολη στιγμή. Συναδέλφισες και συνάδελφοι. Ήθιστε στην Πολωνία να εκφωνούμε το προσκλητήριο των νεκρών ώστε να παραμείνουν στη μνήμη μας ε, πολύ περισσότερο και καλύτερα. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμά όλους τους παρόντες εκ μέρους ε, όλων των Πολωνών. Στην αίθουσα ε, δίνει σήμερα το παρόν σύσσωμη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωποι των κοινοτικών θεσμικών οργάνων, εκπρόσωποι των κρατών μελών, πρέσβης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όπως φαίνεται όλοι χρειαζόμαστε την ενότητα. Εν τη ισχύς, από εκεί αντιλούμε τις δυνάμεις μας. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωρίζουμε ποια είναι η ισχύση, η τεράστια ισχύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε σε αυτήν ακράδαντα. Και οι τελευταίες μέρες μας υπενθύμησαν για μια ακόμη φορά πόσο σημαντική είναι αυτή η ενότητα και η δύναμη. Λεχ Kaczyński. Ε, μαχητής της ε, Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, μέλος της Αλληλεγγύης και αντιπρόεδρος ε, της Αλληλεγγύης κατόπιν πρόεδρος του ΥΠΑ του Ελεκτικού Συμβουλίου. Υπήρξε υπουργός δικαιοσύνης στην κυβέρνηση που Ήμουν εγώ πρωθυπουργό και κατόπιν δήμαρχο της Βαρσοβίας από το 2005 ήταν πρόεδρος της Πολωνική Δημοκρατίας. Μαρία Κατσίνσκα, πρώτη κυρία της Πολωνικής Δημοκρατίας. Ρίσαρτ Κατσορόφσκι, τελευταίος ενεξορία πρόεδρος της Πολωνικής ε, Δημοκρατίας στο Λονδίνο. Και έδωσε τη σκητάλη της εξουσίας στο Λέχ Βαλέσσα τον ε, νεκλεγέντα πρόεδρο. Άννα Βαλεντινόβιτς. Κορυφαία μαχήτρια της αντιπολίτευσης ε, σημαντική μαχήτρια στα ναυπηγεία του και Μετά τη δική της απόλυση από τα ναυπηγεία του Γκτάνσκ ξεκίνησαν οι απεργίες του 1980 που κατέληξαν στην ίδρυση της αλληλεγγύης. Ξίστοφ Πούτρα αντιπρόεδρος της Γερουσίας, πρώην αντιπρόεδρος της ε, Βουλής, μέλος του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη. Γκραζίνα Γκενσίτσκα, πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Νόμου και Δικαιοσύνη, πρώην Υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Υφυπουργός Απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής. Ψεμίσου Αφγκοσεύσκη, αντιπρόεδρος της, του νόμου και της δικαιοσύνης, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη. Αλεξάνδρα Νάταλη Σβιάτ, βουλευτής και αντιπρόεδρος του Νόμου και Δικαιοσύνη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημοσίων Οικονομικών. Σμπίγνιεφ Βάσερμαν, βουλευτής του Νόμου και Δικαιοσύνη, πρώην Υπουργός Συντονιστή σε θέματα ειδικών υπηρεσιών, υπηρεσιών ασφάλειας και πρώην υφυπουργό δικαιοσύνης. Γιανίνα Φετλίνσκα, γερουσιαστής του νόμου και δικαιοσύνη, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας. Στανίσουαφ Ζάιοντς, γερουσιαστής του νόμου και δικαιοσύνη, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας, πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής, συνήγορος υπεράσπισης σε πολιτικές δίκες πριν το 1989. Κριστίνα Μποχένακ αντιπρόεδρος της Γερουσίας οργάνωσε ε, εθνικές ε, κοινωνικές ε, και ε, δράσεις στη δημοσιογραφία πλατφόρμα των πολιτών. Ξέγκος Ντόλνιακ ήταν βουλευτής για τρεις διαδοχικές θητείες πρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών ε, Υποθέσεων, αντιπρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας της Πλατφόρμας των Πολιτών, επικεφαλής εκλογικού επιτελείου της Πλατφόρμας των Πολιτών πριν τις τελευταίες ευρωεκλογέ. Μάτσεϊ Πουαζίνσκι, βουλευτής για τρεις θητείες, πρόεδρος ε, του Σωματείου Πολωνική Κοινότητα πρώην πρόεδρος της Βουλής, πρώην αντιπρόεδρος της Γερουσίας, ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Πλατφόρμας των Πολιτών και περιφερειάρχης στο ΚΝΤΑΝΣΚ. Αρκάδιος Ριμπίτσκι, βουλευτής σε δύο θητείες ε, της Πλατφόρμας των Πολιτών, πρώην Υφυπουργός Πολιτισμού, ε, συνέταξε τα 21 περιακά μανιφέστα της απεργίας ε, των αυπηγείων του Κτάνσκ το 1980 που προηγήθηκαν της ίδρυσης της αλληλεγγύης. Σεμπάστιαν Καρπίνιουκ, βουλευτής της Πλατφόρμας των Πολιτών, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Συνταγματικής Ευθύνης, γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλατφόρμας των Πολιτών, πρώην αντιπρόεδρος, αντιδήμαρχος της πόλης Κοουόμπζεγκ. Γέζη Σμαϊτζίνσκι, Αντιπρόεδρος της Βουλής, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αντιπρόεδρος ε, του Συνδέσμου Δημοκρατικής Αριστεράς και υποψήφιος του κόμματος αυτού για τις προεδρικές εκλογές του 2010. Ιζαμπέλα Γιαρούγκα Νοβάτσκα, βουλευτής στο Σύνδεσμο Δημοκρατικής Αριστεράς, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός κοινωνικής πολιτικής και κυβερνητική εκπρόσωπος στα θέματα ισότητας ευκαιριών ανδρών και γυναικών και πρόεδρος της ε, Ένωσης για την Απασχόληση. Γιολάντα Σιμάνεκ Εκτέρες, βουλευτής ε, του Συνδέσμου Δημοκρατικής Αριστεράς, αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώην επικεφαλής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου Αλεξάνδρ Κβασνιεύσκη και αντιπρόεδρος ε, του κόμματος του Συνδέσμου Δημοκρατικής Αριστεράς. Leszek. Λέσσακ Ντεπτούα. Βουλευτής για δύο θητείες του ΠΕΣΕΛ, του Πολωνικού Λαϊκού Κόμματος. Περιφερειάρχης στην περιοχή Ποτκαρπάτσκι. Ήταν μέλος του ΥΠΑ του Συμβουλίου του Πολωνικού Λαϊκού Κόμματος. Βιεσουαφ Βόντα, βουλευτής του ΠΕΣΕΛ για πρώτη φορά στο Κοινοβούλιο από το 1989. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Μέλος του Συμβουλίου Πολιτικής Προστασίας, Περιφερειάρχης του Τάρνοφ και μέλος του ΕΠΑ του Συμβουλίου, του PSL. Έντβαρτ Βόιτας βουλευτής του ΠΕΣΕΛ για δύο κοινοβουλευτικές θητείες. Πρώην περιφερειάρχης, δήμαρχος του Λουμπέλ, θα ήταν ο 51ος Πολωνός Ευρωβουλευτής στην Ευρωπαϊκή Βουλή μετά την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Βουαντίσουαφ Στάσακ, επικεφαλής του Ιδιαίτερου Γραφείου του Προέδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας, πρώην ε, Υπουργός Ασωτερικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, πρώην Δήμαρχος της Βασοβίας, πρώην μαχητής ε, στην, ε, στο Ανεξάρτητο Σωματείο Φοιτητών. Αλεξάνδρες Σίγκουο, επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Μάριος Χάνσλικ, πρόεδρος, παρά το πρόεδρο της Πολωνικής Δημοκρατίας, υπουργό, συγγνώμη, στο γραφείο του πρόεδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας, Παύε Βίπιχ υπουργό στο γραφείο του Πρόεδρου της Πολωνικής Δημοκρατίας. Στανίσο Βιέζη Κομορόσκι, υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, πρώην υφυπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, πρώην πρέσβης της Πολωνικής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρώην πρέσβης της Πολωνικής Δημοκρατίας στην, στις κάτω χώρες. Άντζεϊ Κρέμερ, υφυπουργό Εξωτερικών. Τόμας Μέρτα, υφυπουργό Πολιτισμού και Εθνικής Κληρονομιάς. Κορυφαίος συντηρητής πολιτιστικής κληρονομιάς. Μάριος Καζάνα, Διευθυντής του Διπλωματικού Πρωτοκόλου του Υπουργείου Εξωτερικών. Σλαβόμιρ Σκρίπεκ. Σλαβόμιρ Σκρίπεκ, πρόεδρος της Πολωνικής Εθνικής Τράπεζας, Κεντρικής Τράπεζας, πρώην αντιδήμαρχος της Βαρσοβίας, μαχητής της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, μέλος ε, Αντικομμουνιστικής ε, οργάνωσης νεολαίας, οργανωτής ε, απεργιών φοιτητών. Καλός σύντροφος. Γιάννος Κοχανόφσκι, δικηγόρος, συνήγορος του πολίτη. Πιότρ Νουρόφσκι, ο επικεφαλής της Πολωνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, επιχειρηματίας, έμπειρος Πολωνός διπλωμάτης. Είμαστε μαζί με την οικογένειά τους αυτές τις δύσκολες στιγμές. Άντζεϊ Ψεβόσνικ, υπουργό εδώ και 17 χρόνια, Γραμματέα ε, γραμματέας ε, του Συμβουλίου Προστασίας της Μνήμης και του Αγώνα. Ήθελα να συμμετάσχει σε αυτή την επιμνημόσυνη τελετή για το ΚΑΤΗΝ και συμμετείχε και στην οργάνωση της έκθεσης για το ΚΑΤΗΝ που λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στανίσου Αφμίκε, δικηγόρος, πρώην ε, δικαστής στο Ανάτοτο Δικαστήριο, αντιπρόεδρος ε, του Συμβουλίου Προστασίας της Μνήμης και του Αγώνα. Δόκτωρ Γιάννος Κουρτίκα, πρόεδρος του Ινστιτούτου Εθνικής Μνήμης. Γιάννος Κρούψκι, ο επικεφαλής του Γραφείου για θέματα μαχητών και άνθρωπων που έχουν υποστεί καταπίεση από το καθεστώς. Υπέστη πολλές διώξεις ε, από τις υπηρεσίες ασφαλείας του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ιωάννα Αγκάτσκα Ιντέτσκα, δικηγόρος, πρόεδρος του Πολωνικού Δικηγορικού Συλλόγου. Στρατηγός Φραντσίσεκ Γκόγκορ, ο αρχηγός του πολωνικού στρατού, ξηράς. Στρατηγός Μπρονίσοφ Κριατκόφσκι, αρχηγός των ειδικών δυνάμεων ασφαλείας του πολωνικού στρατού. στρατηγός Αντζέι Μποάσικ, πτέραρχος μάλλον, αρχηγός των εναέριων δυνάμεων της Πολωνίας, της πολωνικής αεροπορίας. Ταξίαρχος Ταδέος Μποκ, αρχηγός του στρατού Ξηράς. Ταξίαρχος Βοτζίμιος Ποτασίνσκι, αρχηγός των ειδικών δυνάμεων. Αντινάβαρχος Αντζέι Καρβέτα, αρχηγός του πολεμικού πολωνικού ναυτικού. Ταξίαρχος Καζίμες Γκυλάρσκι, ο επικεφαλής της Φρουράς της Βαρσοβίας. Generalmajor, Bischof. επίσκοπος με το βαθμό στρατηγού Σταντέους Πόσκι. επίσκοπος των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Συνταγματάρχης Αρχιεπίσκοπος Μύρον Χοντακόφσκι. der polnischen Oberst Pastor Adam Pilch. Ιερέας Άνταμ Πίρχη. Ευαγγελικός ιερωμένος των πολωνικών ενόπλων ε, δυνάμεων της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Πάτερ Ιαν Οσίσκι, καθολικός ιερωμένος των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων. Πάτερ Roman Πατήρ Ρόμαν Γιέτσις, γερωμένος ε, παρά το πρόεδρο της Δημοκρατίας της Πολωνίας. Καθηγητή Καθηγητής ε, και γερωμένος Ρίτσαρτ Ρουμιάνεκ, πρίτανης ε, του Πανεπιστημίου Βιτσίνσκι της Βαρσοβίας. Πατήρ Μπρόνισλαβ Γκοστόμσκι, εκπρόσωπος της Ένωσης των Οικογενειών του Κατίν. Πατήρ Ιώζεφ Γιόνιτς, εκπρόσωπος της Ένωσης Παραφιάντα. Πατήρ Ζδίσλαφ Κρόλ, εκπρόσωπος της Ένωσης Οικογένειες του Κατίν. Πατήρ Αντζέι Κβάσνικ, εκπρόσωπος της Ένωσης Οικογένειες του Κατίν. Ετβάρτ Ντουχνόφσκι, πρόεδρος της Ένωσης των Θυμάτων της Σιβηρίας. Αντζέι Ζάριος Σκόμσκι, πρόεδρος της Ένωσης των Οικογενειών του Κατίν. και για τα θύματα των οικογενειών του Κατίν, Ταντέους Λουντεμπόφσκι, Άννα Μαρία Μπρόφσκα, Μπάρτος Μπορόφσκι. Μπρονισιάβα, Μπορεύτς, Κράβιετς, Λόφλερ. Καταζίνα Πισκόρσκα. Wojciech Severin. Leszek Solski. Gabriela Sich. Czesław Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συνδέσμου των Στρατιωτών του Εθνικού Στρατού. Στέφαν Μέλακ, πρόεδρος της Επιτροπής του Κατίν. Ζενόνα Μαμοντόβιτς Βόγεκ, συνειδήτρη του Συνδέσμου Οικογενειών του Κατίν. Τερέζα Βαλέσκα Ψιακόφσκα, πρόεδρος του Ιδρύματος Γολγοθάς στην Ανατολή. Εύα Μπονκόφσκα, εγγονή του Μετζουσλάβα Σμοραβίσκη, που, στρατηγού που δολοφονήθηκε στο Κατίν. Σπίγνιεφ Τέμσκι, ε, βετεράνος της εξέγερσης της ε, Βαρσοβίας ε, και τιμήθηκε με, το, με την ύψιστη στρατιωτική διάκριση. Μισλάβ Κομονόφσκι ε, τιμήθηκε επίση με την ύψιστη στρατιωτική, στρατιωτική τιμή. τη μιλιτάρη. Janjana Νατουσιέβιτς Miller, Überlebende eines Lagers in Sibirien επιζών ενός στρατοπέδου στη Σιβηρία. Janusz Zakrzniewski, Schauspieler. Ηθοποιός. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Οι συνεργάτες του Προέδρου της Δημοκρατίας της ε, Πολωνίας, Καταζίνα Δαβαζίνσκα. Ο Αλεξάνδρ Φεντόροβιτς. Dariusz Jankowski. Oberst Dr. Wojciech Lubinski. Γιατρός Lubinski, Wojciech Lubinski. Barbara Maminska. Isabella Tomaszewska. Lieutenant Colonel Jaroslav Flosiak. Αντισυνταγματάρχης Γιάροσλαφ Φλόσακ. Captain Darius Mikawowski. Κυβερνήτης Darius Misalowski. Η Πολοχαγός Πάβελ Γιάννησεκ. second lieutenant Piotr. Ανθιπολογαγός Πάβελ Νόσεκ, Πιότρ Νόσεκ, συγγνώμη. Warrant officer Arthur Francis. Αξιωματικός Arthur Francis. Αξιωματικός Πάβελ Κραζένσκι. Warrant Officer Jacek Surówka. Αξιωματικός Jacek Surówka. Warrant Officer Αξιωματικός Marek Ulerik. Junior Warrant Officer Agnieszka. Υπαξιωματικός Agnieszka Pokrutka Wyslawek. Τα μέλη του πληρώματος. Πιλότος Ακάβιτ Προτάσεκ, πιλότος, κυβερνήτης μάλλον της πτήσης. Ρόμπερτ Κρίσνα, πιλότος. Υπολογός Άρτος Διέτεκ. Αξιωματικός Αντρέη Μισάλακ. Νατάλια Γινούσκο. Μπάρμπαρα Ματσέιτσικ. Ιουστίνα Μουνιούσκου